Ας συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το σύστημα ακριβώς ε, των, ε, της ετικετοποίησης ε, όσον αφορά τις άμεσες ε, πωλήσει ε, τοπικής ε, παραγωγής γεωργίας και έκθεση της Επιτροπής για την, τα, προϊόντα με την εισαγωγή ένδειξης προϊόν ισιωτικής γεωργίας ως προαιρετικής ένδειξης ποιότητας. Αυτές οι δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν όπως προαναφέρθηκε θα μας απασχολήσουν, διότι κατατέθηκαν μετά από αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά την ποιότητα γεωργικών προϊόντων. Η πρώτη έκθεση αφορά την τοπική γεωργία και τις άμεσες πωλήσει. Η δεύτερη αφορά ρυθμίσεις ε, του όρου ποιότητας, ε, ποιοτικής, ε, ποιοτικού προϊόντος όσον αφορά την ισιωτική γεωργία. Για την πρώτη έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει αν αυτή η πρωτοβουλία δίνει την βέλτιστη εναλλακτική δυνατότητα ώστε να χρησιμοποιούνται όροι ποιότητας που θα χρησιμοποιούνται εθελοντικά. Και στην δεύτερη έκθεση επεξηγεί τα υπέρ και τα κατά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ενδυνάμει χρήσης ε, της ένδειξης προϊόντος ε, νησιωτικής γεωργίας. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι έχουμε το θέμα της παραγωγής. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας επεξηγήσει περί τίνος πρόκειται πρώτα απ' όλα. Και σύμφωνα με τις σημειώσεις μου, ο κύριος Έλχαρντ θα λάβει τον λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να καλωσορίσω και τους άλλους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που πρέπει να γίνει, καθώς επίσης και τους φιλοξενουμένους που έχουμε εδώ παρόντες απόψε ανάμεσά μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι Κύριε Έρχαντ, έχετε τον λόγο από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καταρχήν θα ήθελα πρώτα απ' όλα να παρουσιάσω την έκθεση της Επιτροπής ε, για την ε, επισήμανση για τα προϊόντα τοπικής ε, γεωργίας και τις άμεσες πωλήσει. Και αμέσως μετά στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τα, την έκθεση για τα νησιωτικά προϊόντα, προϊόντα νησιωτικής γεωργίας. Ο κανονισμός λοιπόν για ποιοτικές ε, ε ενδείξεις ε, όπως ε, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση αν μια νέα ρύθμιση για τέτοιου είδους προϊόντα για την τοπική γεωργία και τις άμεσες πωλήσει θα έπρεπε να εισαχθεί με τέτοιου είδους ε, ε, καθοριστικά ε, στοιχεία ώστε να υποστηριχθεί η πώληση και διάθεση αυτών των τοπικών προϊόντων. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επίσης κριτήρια όπως π.χ. η δυνατότητα ε, όσον αφορά την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα κατά την αλυσίδα ε, αγοράς και πώλησης αυτών των προϊόντων να την μειώσουμε, να μειώσουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Για να δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει έκανε πολυσχηδείς δραστηριότητες ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και διαβουλεύτηκε με τα κράτη-μέλη και τους εκπροσώπους τους είχε ε, συμπόσια, ημερίδες μελετών, σεμινάρια τα οποία διεξήγαγε κτλ. Η εξέλιξη των άμεσων πωλήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωστάτ μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετική, υπέχει πολύ διαφορετικά στοιχεία. Όσον αφορά τους καταναλωτές, οι μελέτες δείχνουν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για την αγορά τοπικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων από την τοπική γεωργία. Τώρα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δηλαδή τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την άμεση πώληση σε σχέση με την τοπική γεωργία τέτοιων προϊόντων και τις επιπτώσεις ε, στην τοπική οικονομία. Ανέλησε μελέτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν ε, οι σχέσεις μεταξύ της ε, αλυσίδας προϊόντων και των, της κάλυψης των αναγκών και μείωση, μείωση των ε, της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος για να μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα αυτά τα στοιχεία. Μικρές αλυσίδες δείχνουν οι μελέτες ε, στην πώληση τέτοιων προϊόντων έχουν θετικές επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον όταν είναι μικρές οι αποστάσεις. Όταν λειτουργούν δηλαδή τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο και έχουμε εποχικά, εποχικά ε, παραγόμενα προϊόντα και χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες ώστε να έχουμε μικρό ίχνος διοξιδίου του άνθρακα, μικρό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις ότι άμεση τοπική πώληση αυτών των προϊόντων γενικά έχουν, έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό δεν ισχύει. Πολύ περισσότερο μια ολόκληρη σειρά όρων και προϋποθέσεων πρέπει να τηρούνται και να ισχύουν για να υπάρχει αυτό το θετικό στο περιβάλλον αποτέλεσμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σε μεγάλο βαθμό, ε, διαβουλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό με πολλούς ε, επαΐοντες ώστε να μπορέσει να ε, διαγνώσει ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για ένα τέτοιο λειτουργικό σύστημα. Συμφώνησαν οι επαΐοντες ότι ένα πιθανό τέτοιο σύστημα θα πρέπει εθελοντικής φύσης να είναι και όχι υποχρεωτικού χαρακτήρα και ότι η πιστοποίηση και η αδειοδότηση θα πρέπει να αποφεύγονται διότι επιβαρύνουν και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες και δημιουργούν γραφειοκρατική επιβάρυνση και θα πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια για την ένταξη τέτοιων προϊόντων στο πλαίσιο αυτό. Οι επαΐοντες που διαβουλεύτηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσαν επίσης ότι ένα σύστημα ε, σήμανσης είναι μόνο τότε σκόπιμο όταν συνδυάζεται με άλλα μέτρα ή συμπληρωματικά λειτουργεί με άλλα μέτρα ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να υποστηριχθούν στην αναζήτηση εναλλακτικών δυνατοτήτων. Τέτοια μέτρα υφίστανται στην ανάπτυξη του χώρου της υπαίθρου για παράδειγμα. Συμβουλευτικές ε, διαδικασίες, ε, υποστηρικτικές διαδικασίες ε, για την εξέλιξη της διοχέτευσης και διάθεσης προϊόντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν παράλληλα με, μια, με ένα αυθύπαρκτο αυτόνομο τέτοιο σύστημα επισήμανσης ανέλησε κατά πόσον μια εθελοντική ποιοτική ένδειξη μπορεί να αναφέρεται σε αυτό το πλαίσιο και κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να ήταν μια λύση εθελοντικές ποιοτικές ενδείξεις. Είναι ένα νέο σύστημα ποιοτικών αναφορών που με τις, τις εισαγωγές ποιοτικών χαρακτηριστικών μπορεί να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα το ε, μια τέτοια ένδειξη είναι προϊόν ορεινής γεωργίας, για παράδειγμα. Berg Product. Σύμφωνα με τις ε, μελέτες επιπτώσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέτοιες ποιοτικές ενδείξεις, οι εθελούς, εθελοντικού χαρακτήρα τέτοιες ε, ενδείξεις ε, είναι ένα, μια δυνατότητα να καταδείξουν οι γεωργοί κατά πόσον στην μεταποίηση υπήρξε πρόσθετη προσπάθεια από πλευρά του ώστε να μπορέσει να αντισταθμιστεί από πλευρά τιμή προϊόντος ε, η προσπάθεια αυτή. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτές τις μελέτες τη ποιο είναι. Είναι ότι καταρχήν υφίσταται ανάγκη για πραγματικά αυθεντικά προϊόντα, γεωργικά προϊόντα που θα μπορούν σε μικρές αλυσίδες να διατίθενται στην αγορά, ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν ότι είναι μικρής απόστασης διαφο ε, ε, αποστάσεις που καλύπτονται. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για αυτά τα θέματα. Η ανάπτυξη της αλυσίδας αυτής συναρτάται με, την αντιμετώπιση πάρα πολλών προκλήσεων για τις οποίες πρέπει να αναζητηθεί άλλη δυνατότητα επίλυσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα επίπεδο κρατών μελών υπάρχουν τέτοια μέσα τα οποία όμως ε, δεν είναι ευθύ εκ προημίου τα πιο ενδεδειγμένα. Μια νέα ετικέτα για παράδειγμα που θα εισαχθεί θα μπορεί να απλουστεύσει τον χαρακτηρισμό αυτών των προϊόντων. Δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιβάρυνση και θα πρέπει να διασφαλίζει την νομική βεβαιότητα για τους καταναλωτές ότι αγοράζουν αυτό που επιθυμούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει την έκθεσή της με διαφορετικά ερωτήματα που θέτει, διαφορετικά ζητήματα τα οποία θέτει η προσυζήτηση, ώστε αυτή η έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο <coughs> και από πλευράς του Συμβουλίου να διευκολυνθεί. Το πρώτο ερώτημα είναι αν τα διαφορετικά, διάφορα μέσα τα και εργαλεία που υπάρχουν ήδη σήμερα στο, επί, στο κοινοτικό επίπεδο για την προαγωγή της τοπικής γεωργίας και την προώθηση των άμεσων πωλήσεων είναι τα ενδεδειγμένα και τα πιο κατάλληλα. Δεύτερο ερώτημα. Μια και ολόκληρη σειρά, μια ολόκληρη σειρά ομάδων και συλλόγων συμφερόντων έχουν καθοριστεί που για παράδειγμα σε σχέση με τη σύναψη συμβάσεων ή ε, ε, συμβολέων για την ε, ανάπτυξη των τοπικών πολίσεων θα πρέπει να εξεταστούν. Εδώ πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διατάξεις που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπεριέχουν ένα βαθμό ελαστικότητας που όμως δεν τον εξαντλούμε πλήρως όπως θα έπρεπε. Το ερώτημα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τι πιστεύουν. Συμμερίζονται αυτή την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όχι. Ή μήπως στο κοινοτικό επίπεδο θα έπρεπε να υπάρχουν πιο, πιο σαφείς ενδείξεις για τις διατάξεις ε, για την διάθεση ε, άμεση πώληση τέτοιων προϊόντων. Περαιτέρω υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα μια και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν ήδη διατάξεις ε, για την ε, ε, ετικετοποίηση και επισήμανση τέτοιων προϊόντων, τίθεται το ερώτημα αν χρειαζόμαστε μια νέα ρύθμιση, αν αυτή θα προσφέρει κάτι καινούριο στους γεωργούς ως κέρδος και αν θα συνεισφέρει ώστε οι καταναλωτές να έχουν πληροφορίες στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε σχέση με τις άλλες ετικέτες. Μια τέτοια ετικετοποίηση τι θα είναι, ένα λογότυπο, ένα σύμβολο, θα εμπεριέχεται ή όχι σε μια τέτοια ετικετοποίηση. Και τέλος και το ερώτημα το οποίο τίθεται Πώς μπορεί κανείς μια τέτοια ευρωπαϊκή ρύθμιση να την δημιουργήσει και να την εκπονήσει ώστε να μην επιβαρύνονται οι γεωργοί με περιττές επιβαρύνσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται επαρκώς τα συμφέροντα των καταναλωτών με εχέγγυα που θα τους προσφέρονται. Αυτή είναι μια σύντομη λοιπόν παρουσίαση από πλευράς μου αυτής της έκθεσης. Και ολοκληρώνω έτσι για την ε, άμεση τοπική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και την διάθεσή τους στην αγορά με τοπικές πωλήσει. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση για τα προϊόντα, προϊόντα νησιωτικής γεωργίας, θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής. Και εδώ πάλι έχουμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνταχθεί μια έκθεση από πλευράς μας. Αν μια νέα ένδειξη, μια νέα αναφορά προϊόν νησιωτικής γεωργίας πρέπει να εισαχθεί ή όχι, προαιρετικά ως ένδειξη ποιότητας. Και εδώ πρέπει πάλι να λάβουμε υπόψη ότι η συγκεκριμένη εντολή που μας δόθηκε είναι αυτό να εξεταστεί υπό το πλαίσιο μιας εθελοντικής ποιοτικής ένδειξης και όχι μέσα στο πλαίσιο μιας υποχρεωτικής ένδειξης από πλευράς ετικετών. Από την άλλη πλευρά θα έπρεπε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επακριβώς κατά πόσον είναι ενδιαφέρον για τέτοιου είδους προϊόντα που στοχεύουν στην ε, ανθρώπινη κατανάλωση και κατά πόσον αυτά μπορούν να προαχθούν εφόσον οι πρώτες ύλες για την παραγωγή αυτών των προϊόντων προέρχονται από νησιωτικές περιοχές και σε περίπτωση μεταποίησης πρέπει πάλι και η μεταποίηση να διεξάγεται, να ολοκληρώνεται στις νησιωτικές περιοχές για να θεωρούνται νησιωτικά, προϊόντα νησιωτικής γεωργίας. Αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να απαντηθούν. Ευθύ εξ αρχή στο έργο τη είδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο ορισμό αυτού που είναι νήσος το τι είναι νήσος είναι διαφορετική, χάνει διαφορετικής ερμηνείας ανάλογα με το στόχο του ορισμού. Σε ενωτικό επίπεδο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις διορισμού νήσων. Η ίδια η έκθεση εδώ δεν καταλήγει σε μια καθοριστική τελεσίδικη απόφαση ή επιλογή μεταξύ αυτών των ορισμών. Η έκθεση καταδεικνύει ότι η νησιωτική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια ολόκληρη σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων. Από πλευράς προϊόντων τώρα που εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νησιωτικής Γεωργίας βλέπουμε ότι οι νησιωτικές εκμεταλλεύσεις στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεγαλύτερο μέρος αφορούν κυπευτικά προϊόντα Η νησιωτική γεωργία έχει ένα χαρακτηριστικό και αυτό έπρεπε να αναλύσουμε έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η νησιωτική γεωργία που κυρίως ανταποκρίνονται σε διαρθρωτικά προβλήματα και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και δεν αναφέρονται τόσο πολύ στα χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων. Δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυπικά τέτοια χαρακτηριστικά νησιωτικού χαρακτήρα να ταυτοποιήσει που θα μπορούσαν να, να αποτελούν ας πούμε ένα συμπέρασμα αυτών των μελετών. Και περαιτέρω τι δείχνει. Καταδεικνύει η έκθεση ότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά προϊόντων που ήδη έχουν μια αναφορά γίνεται μία αναφορά στην νησιωτική τους προέλευση και την νησιωτική διάθεση στο εμπόριο. Όμως γενικά ο όρος νησιωτικός δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά. Πιο συχνά χρησιμοποιείται το όνομα του αρχιπελάγους ή της ε, νησιωτικής συστάδας, ε, γιατί ίσως αυτό είναι καλύτερα ενδεδειγμένο για την ε, καλύτερη εμπορία, διάθεση στο εμπόριο αυτών των προϊόντων. Τώρα, όσον αφορά την πρόσθετη αξία μιας εξειδικευμένης ε, ενωτικής ε, ένδειξης χαρακτηρισμού νησιο, προϊόντος νησιωτικής γεωργίας, οι απόψεις δίστανται ποια είναι η αξία μιας τέτοιας επισήμανσης. Δίστανται και σε μεγάλο βαθμό κιόλας στην διάθεση στην εμπορία αυτών των προϊόντων η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών αναφέρουν τις ε, νήσους που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά στην παραγωγή ενός προϊόντος και έτσι υπό αυτό το πλαίσιο γίνεται μια αναφορά μιας νήσου. Δεν μπορέσαμε να βρούμε μια μάρκα ή ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που να συνενώνουν όλες τις νήσους ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους και γεωγραφική τους ε, ένταξη. Οριζόν οριζόντια λοιπόν εγκάρσια μόνο για μικρά νησιά ή μια, ένα, κάποια μικρά δανέζικα νησιά ή στη Φινλανδία χρησιμοποιούνται τέτοιες ενδείξεις. Διότι κατά τα άλλα πάντα μια συγκεκριμένη νήσος αναφέρεται πάντα με το όνομά της και επιπλέον διαπίστωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους διάφορα νησιά και η αναφορά σε ένα συγκεκριμένο νησί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει το προϊόν αυτής της νήσου να αποκτήσει ταυτότητα ξεχωριστή στην αγορά. Τώρα, όσον αφορά τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της εισαγωγής μιας εθελοντικής ένδειξης ποιότητας ή αναφοράς ποιότητας όσον αφορά προϊόν ισιωτικής γεωργίας, η έκθεση αυτή απαριθμεί τα εξής στοιχεία ένα προς ένα. Ένα επιχείρημα για μια τέτοια εθελοντική ε, ποιοτική ένδειξη θα ήταν και είναι ότι οι ποιοτικέ τέτοιε εθελοντικέ ενδείξει με πολύ μικρή γραφειοκρατική ε, επιβάρυνση και πολύ μικρή ε, επιβάρυνση για ελέγχου ή εποπτεία συνδέεται. Ιδιαίτερα για μικρο, μικρούς παραγωγείς σε μικρά νησιά θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είναι ενδιαφέρον ως προοπτική. Αν δεν έχουν επαρκή, επαρκή επαρκή διάσταση επαρκώς μεγάλη διάσταση αυτές οι εκμεταλλεύσεις ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν άλλου είδους ε, ε, ενδείξεις. Αρνητικά στοιχεία, μεταξύ των αρνητικών στοιχείων για την χρήση η δημιουργία μιας νέας εθελοντικής τέτοιας ένδειξης νησιωτικών προϊόντων απαριθμεί έκθεση για παράδειγμα ότι μια τέτοια ένδειξη θα μπορούσε να, είναι αρνητική, να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς εκείνους που χρησιμοποιούν ήδη κάποιες, ε, κάποιους χαρακτηρισμούς ή κάποιες, κάποια στοιχεία ε, διαφοροποίησης σε σχέση με τα προϊόντα τους. Εδώ θα υπήρχε για παράδειγμα η, ε, ο κίνδυνος διαφοροποίησης ιστορικά χρησιμοποιούμενων όρων Επιπλέον, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια γενική ε, κάλυψη με τέτοιους ε, όρους ε, ή ενδείξεις για νησιωτικά προϊόντα. Ο όρος νήσος δεν επαρκεί για να χαρακτηρίζονται τέτοια προϊόντα όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, τα περισσότερα νησιωτικά προϊόντα δεν εξάγονται όλα, αλλά καταναλώνονται τοπικά ή διατίθενται στην υπηρετική τους ε, ε, ενδοχώρα και γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο στο επίπεδο των κρατών μελών να υπάρξει μια τέτοια αρρύθμιση, των κρατών μελών στα οποία διοχετεύονται αυτά τα νησιωτικά προϊόντα προς κατανάλωση. Στο τέλος τέλος το εύρος των προϊόντων που για τέτοιου είδους ε, ποιοτικέ ενδείξεις θα μπορούσαν να εξεταστούν λόγω του περιορισμού των πρώτων υλών από, με, με νησιωτική προέλευση και λόγω των ε, περιορισμών που συνεπάγονται από τις ε, συνθήκες συνθήκες έχουν ένα πολύ περιορισμένο εύρος ως εμβέλεια και τα διαθωτικά προβλήματα των νησιών θα μπορούσαν ίσως καλύτερα να αντιμετωπιστούν με τα σημερινά διαρθρωτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και όχι τόσο με μια προσπάθεια ετικετοποίησης ή διαφοροποίησης μέσω ετικετα, ετικέτας ή συσκευασίας. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτών των μελετών και τα οποία έχει συντάξει στην έκθεση αυτή για τα νησιωτικής προέλευσης προϊόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μία ομάδα επισκεπτών από νέους εκπροσώπους γεωργών και μελλοντικών γεωργών. Μόλις ήρθαν. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω από ποια χώρα οι χώρες βρίσκονται, έχουν έρθει, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Ήθελα να σας το πω όμως αυτό ότι είναι εδώ μαζί μα. και τώρα πάμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την παρέμβαση της Κομισιόν. Ο πρώτο που θα πάρει το λόγο, Ποιο είναι? Α, οι επισκέπτε είναι από την Ιταλία. Είναι κρίμα που δεν είναι εδώ ο κύριο Δεκάστρο για να σα ε, καλωσορίσει. Εν πάση περιπτώσει, οι ευρωβουλευτέ τώρα έχουν τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Ανδρεού. Ευχαριστώ τον εισηγητή της Κομισιόν για όσα είπε στην παρουσίαση του. Παρότι δεν κατάλαβα απόλυτα όλα τα στοιχεία, γιατί δεν είμαι και πολύ παλιό στο κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω πού το πάει η έκθεση. Ακριβώς. Κατάλαβα τη διαδικασία όμως. Πάντως ε, συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα υποβάλει μια έκθεση πρωτοβουλίας για τα θέματα του εδαφικού σήματος. Και πολλά από τα σημεία που εμπεριείχε η έκθεσή μου τα άκουσα σήμερα, άκουσα όρους από την Κομισιόν για την ετικετοθεσία, η οποία θα έχει ένα μεταφικό χαρακτήρα τελικά. Αν η δική μου έκθεση πρωτοβουλία επέτρεψε στην Κομισιόν να αντιδράσει τόσο γρήγορα και να λάβει υπόψη το θέμα τη εδαφικότητα, χαίρομαι ιδιαίτερω. Μια και η Κομισιόν ούτω ή άλλω είχε εκφράσει κάποιε επιφυλάξει. Οπότε, Πολλές φορές έχει εκφράσει αντιρρήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, οπότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Πάντως, σήμερα το απόγευμα ακούστηκαν διάφορα θέματα που βρίσκουν σύμφωνο. Τίθεται το ερώτημα που είχα θέσει και εγώ στην έκθεσή μου, της ε, κυκλικής οικονομίας. Το πρόβλημα της ε, οριζόντιας ε, λειτουργίας της γεωργίας και πώς μπορούμε οι διάφοροι φορείς να αλληλεπιδράσουν, ώστε να δημιουργήσουμε πραγματική προστιθέμενη αξία. Να υπάρξει αυτή η παραγωγή η εντόπια και να έρθει σε επαφή ο παραγωγός με τον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής να είναι και από τα αστικά κέντρα και από τις περιοχές γύρω από τα αστικά κέντρα. Για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι στη διάθεση της Κομισιόν για να συνεχίσουμε τις εργασίες επί του φακέλου αυτού, γιατί μου φαίνεται πολύ σημαντικό τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, εν ώψη της ε, προετοιμασίας της μεροντικής ε, μεταρρύθμισης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το νέο στοιχείο της εδαφικότητας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πού συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά να μην ξεχάσουμε και πού παράγονται αυτά τα προϊόντα ε, και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα προωθήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν για αυτό το περίπλοκο θέμα τους επόμενους ε, μήνες και χρόνια να ασχοληθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γιάρ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω, ας το πω έτσι, για τον αναστοχαστικό τόνο που εμπνέει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει ερωτήσεις και ερωτήματα μετά την ακρόαση των επαϊόντων και την ενασχόλησή της με το θέμα. Και αυτά τα ερωτήματα είναι ακριβώς τα ουσιοδέστερα ερωτήματα. Για την άμεση διάθεση στην αγορά, οι άμεσες πωλήσει είναι το απλούστερο που μπορεί να κάνει κανείς. Πρέπει πολύ ευαίσθητους μηχανισμούς να χρησιμοποιήσουμε βέβαια και συνετούς μηχανισμούς μέσα στο πλαίσιο της επικουρικότητας και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της ε, του κεντρικού σχεδιασμού από τις Βρυξέλλες πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν με το σωστότερο τρόπο. Να μην καταστραφούν πράγματα όπως για παράδειγμα για τις υγειονομικές διατάξεις ε, σφαγίων που ε, ακούγονται πολύ λογικά. Έχουν δικαίωμα οι καταναλωτές να μπορούν να αγοράζουν ε, τρόφιμα τα οποία θα έχουν παραθεί με τους πιο υγιεινούς τρόπους ε, από πλευράς παραγωγής. Ήθισε στη Γερμανία τα μικρότερα ζώα, λαγί, ε, κουνέλια, ε, γουρουνάκια, οι ίδιοι οι γεωργοί να μπορούν να τα ε, σφάζουν. Σε αυτή τη νέα υγειονομική διάταξη υπήρχε μεγάλη επίπτωση αύξησης επενδύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μονάδες των παραγωγών. Ένα στοιχείο της άμεσης διάθεσης στην αγορά έπαψε να ισχύει. Η άμεση δηλαδή σφαγή των ιδίων των, γεωργών, κτηνοτρόφων αυτών των προϊόντων. Και η άλλη επίπτωση ήταν ακόμα πιο σημαντική. Ήθιστε στον χώρο της, ε, ε, των κτηνοτρόφων να έχουν να κρατούν τέτοια ζώα και να μπορούν να σφάζουν αυτά τα ζώα ανάλογα με την ανάγκη τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους με κρέας και με τις πιο ε, καλές συνθήκες μπορούσαν να το κάνουν αυτό και να τα καταναλώνουν. Τώρα απαγορεύονται όλα αυτά, δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν σφαγεία, προβλέπονται άλλες διαδικασίες ε, και ε, τι συμβαίνει τώρα σε σχέση με τους γεωργούς και κτηνοτρόφους κάτι που είχαμε καλό στόχο να πετύχουμε κάτι καλό με αυτό αν αντέβαινε τη σωστή επίτευξη των στόχων και υπονομεύθηκαν τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές λοιπόν και κάνουμε λόγο εδώ για τις άμεσες πωλήσει. άμεσες πωλήσει πρέπει να δίνουν στον καταναλωτή τα ηχέγγια ότι προέρχονται αυτά τα προϊόντα από την δική του περιοχή, από την ίδια αυτή την περιφέρεια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό όμως το οποίο χαρακτηρίζεται έτσι πράγματι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για παράδειγμα όταν κάποιος παράγει λουκάνικα εντάξει και όταν πρέπει να αγοράζει τα πρώτα, ε, τα, τις πρώτες ύλες καταλήγουμε πολλές φορές σε μεικτά προϊόντα που ε, παράγονται με, την, με χείριο κρέας, ε, με βόηο κρέας και γι' αυτό σε σχέση με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε χαρούμενοι, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας ότι αρχίζει μια συζήτηση αυτών των πραγμάτων που πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία ώστε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των καταναλωτών. Να υπάρχει μια ευκαιρία ώστε με τις άμεσες πωλήσει να υποφελούνται οι καταναλωτές. Πρέπει να μπορούμε να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά το πλαίσιο των άμεσων πωλήσεων και το υπονομεύσουμε. Από την άλλη πλευρά πρέπει να μπορούν σε σχέση με τους καταναλωτές να υλοποιούνται οι στόχοι, να παίρνουν οι καταναλωτές το προϊόν το οποίο επιθυμούν αναβαθμισμένης ποιότητας. Δεν είναι λοιπόν το πιο απλό και δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ωραία. θα πρέπει να αδειάσουμε λίγο χώρο στο, στον καράζ για τα ζώα. Έχουμε επίσης εδώ και Βέλγους δημοσιογράφους, πρέπει να πω. Πάμε τώρα στον επόμενο μιλητή, που είναι ο κύριος Ταραμπέλα. Έχετε το λόγο Ορίστε, ένας Ιταλός θα σας χαιρετήσει, λέει ο πρόεδρος. Συμφωνώ με τον κύριο Αντριέ και τον κύριο Γιάν. Η πρόταση της Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, στην έκθεσή της, πηγαίνει προς μια σωστή κατεύθυνση μαζί και σύμφωνους. Το να διευκολύνουμε την μεταποίηση των προϊόντων στην γεωργική εκμετάλλευση είναι καλό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, αλλά εκεί που θέλουν να το κάνουν θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Γιατί άλλο μεταπίσει άλλο παραγωγή, έτσι. Ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι οι κανόνες, οι οποίοι καμιά φορά είναι εντελώ ακατάλληλοι για τους μικρούς παραγωγούς. Συχνά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, σε θέματα ας πούμε ασφάλειας των τροφίμων, έχουμε κανόνες που δεν είναι καλοί για τους μικρούς. Θα πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν κάποια ευελιξία. Το πρώτο που θέλω να τονίσω, και είναι δύο αυτά που θέλω να τονίσω, είναι το εξή. Για τα μέσα που έχουμε, για τα εργαλεία. Τι θα κάνουμε με αυτή την έκθεση. Συνήθως εξετάζουμε σχέδια οδηγιών ή κανονισμών, είτε εκθέσεις πρωτοβουλία συναδέλφων, όπως έκανε ο Ερίκ Αντριό πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα, να μου πει η Κομισιόν το εξή. Καλή έκθεση τη, ενδιαφέρουσα είναι, αλλά ποιο θα είναι το μέλλον της. Έχουμε στι 25 Μαΐου και τις εκλογές. Μάλλον θα έχουμε, καλά θα έχουμε νέο επίτροπο, αλλά πέρα από αυτό τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτή την έκθεση που μας παρουσίασε η Επιτροπή. Καλό θα ήταν να μας πει. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι το 2014 είναι η ειδική χρονιά. Ε, γεωργική παραγωγή τώρα που συνδέεται με, την, με το έδαφος το οποίο παράγεται. Επίσης, να μου πει η Κομισιόν τι προθέσεις έχει για την ετικετοθεσία. Γιατί δεν θα πρέπει να έχω μια ετικετοθεσία υπερβολική που παραπλανά τον ε, καταναλωτή. Την εξήγηση ότι εννοώ. Όταν μιλάμε για παραγωγή και προέλευση της παραγωγής, παραδείγματος χάρη κοτόπουλων. Φανταστείτε ότι μιλάμε για καταγωγή και όχι προέλευση. Ε, δηλαδή, ε, προέλευση είναι ο, ο τόπος της τελευταίας Αν το κοτόπουλο έρχεται από μία άλλη ήπειρο και βάζουμε λίγα μπαχαρικά, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι που όχι κατά ανάγκη γκαράζ, έτσι. Ε, δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτό το πράγμα τοπικό προϊόν. Υπάρχουν τόσε ετικέτες σήμερα. Μου, θα σας πω ένα παράδειγμα που μου ανέφεραν για την Ιταλία. Ε, μάλιστα μια μεγάλη εταιρεία, Καραπέλη, η οποία ε, θα μετεγκατασταθεί στην Ισπανία. Ε, δεν θα είναι πια Ιταλικό λοιπόν το προϊόν, αλλά Ισπανικό. Μπορεί να ονομαστεί και Καραπελίτος. Δεν θα πρέπει η εδαφική παραγωγή, ε, η παραγωγή των μικρών παραγωγών να αλλοιωθεί από μια ετικέτα που θα είναι τελείως διαφορετική ε, και που παραπλανά τον καταναλωτή. Θα πρέπει ο καταναλωτής, ας πούμε, όταν αγοράζει κοτόπουλα στη φάρμα, να ξέρει ότι εκτράφηκαν εκεί στη φάρμα. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνη. Και σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι οι περιφέρειες που έχουν παραγωγές υψηλή αξίας, παραδείγματο χάρη στα γαλακτοκομικά, έχουν πληγεί λιγότερο από άλλους. Όταν, α πούμε, οι είναι ασταθής. Έχουν λοιπόν μία πηγή εισοδήματο πολύ σταθερή. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι, οι παραγωγοί να προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα. Αλλά προσοχή να μην λένε ψέματα. Και ούτως ώστε και ο Καταναλωτή να έχει εμπιστοσύνη στην ετικέτα. Το σκέφτηκε αυτό η Κομισιόν. Σκέφτηκε αυτό το πρόβλημα της ετικετοθεσίας, που ετικέτες που είναι ασαφείς, που, δεν, που είναι παραπλανητικές, παραδείγματο χάρη ε, ετικέτες που ψεύδονται για την προέλευση του προϊόντος που αγοράζει ο καταναλωτής. Ε, χάρη για το κρέας ή προϊόντα που βασίζονται στο κρέας. Πρόεδρος, Νομίζω ότι καλό θα, καλό θα είναι οι παραγωγοί να μην έχουν να αντιμετωπίσουν υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος ε, στην γεωργική εκμετάλλευση. Ο τελευταίος τώρα ο μιλητής, ο κύριος Βόιτσετσόφσκι. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Γιάρ, ότι υπάρχει πρόβλημα με τα τοπικά σφαγεία, όπου η περιοριστική ευρωπαϊκή νομοθεσία τους εξοβέλσει από την αγορά. Το βλέπουμε αυτό στην Πολωνία. Υπάρχουν περιοχές όπου πρέπει να ταξιδέψεις εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρεις το πιο κοντινό σφαγείο για να παραδώσεις τα ζώα σου. Αυτό το έχουμε συζητήσει. Πριν από κάνα χρόνο, δεν απαντώμε, όταν, απατώμε, όταν μιλήσαμε για μια έκθεση για τη μεταφορά ζώων, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει ότι ήθελε ο χρόνος ε, μεταφοράς των ζώων να είναι το πολύ 8 ώρες. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό δίκτυο σφαγείων. Γιατί το να μεταφέρεις ε, τα ζώα σου σε μεγάλες αποστάσεις, τα επιβαρύνεις, τα κουράζεις και επιπλέον ε, έρχεσαι και αντιμέτωπος με τα δικαιώματα, με τις οργανώσεις δικαιωμάτων των ζώων. Ε, επίσης είναι κακό και για το καταναλωτή. Γιατί κοστίζει και περισσότερο αυτή η μεταφορά. Τότε και η επιβάρηση αυτή μεταφέρει στον τελικό καταναλωτή. Εγώ δεν λέω να σφάζουμε τα ζώα σε ένα γκαράζ όπου να είναι, αλλά θα πρέπει κάποια τοπικά σφαγεία ε, να βρίσκονται κοντά στι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που να έχουν κάποια στάντας, έτσι, που να σέβονται κάποια πρότυπα. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί. Και τώρα, δεύτερο θέμα, η γραφειοκρατία δημιουργεί τέτοια προβλήματα ε, που δεν θα φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της επισήμασης, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα πια για να επισημάνουμε. Ας πούμε στην Πολωνία. Υπήρξαν τόσες αλλαγές που δεν συζητήθηκαν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε, παραδείγματο χάρη, αλλαγές ε, στις, στους τόπους που μπορούμε να καπνίζουμε στην... Συγγνώμη, ε, έχουν αλλάξει οι κανόνες για τα καπνιστά προϊόντα. Άλλαξαν τόσο οι κανόνες που χρειάστηκε να κλείσουν να κάρο ε, ας πούμε μονάδες που κάπνιζαν ε, κρέατα κτλ. Για τυριά. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ετοιμάζεται υποπίεση μεγάλων γεωργικών παραγωγών που δεν καπνίζουν καν το κρέας, αλλά που βάζουν χημικά για να μυρίζει απλώς καπνιστό. Εγώ είχα θέσει και σχετικό ερώτημα στην Κομισιόν και ελπίζω να ακούσω κάποια στιγμή κάποια απάντηση. Πρόεδρος. Τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών. Μετά την πρόσφατη συνάντηση με γεωργούς, θα ήθελα να σας πω και εγώ κάποιους προβληματισμούς μου. Το πρόβλημα που μόλις ακούστηκε είναι πολύ έντονο. Η δυνατότητα σφαγής ε, των ζώων κοντά στην, ε, στον τόπο παραγωγής τους είναι τεράστιο θέμα. Γιατί αν χρειάζεται γιατί αν υπάρχει τέτοιο σφαγείο, τότε μπορεί να σφαγούν εκεί τα ζώα και να πουληθούν και τοπικά. Αλλιώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Πώ θα τα πουλήσει κοντά τα σφάζει ε, χιλιόμετρα μακριά. Ε, υπάρχει και το αστείο. Αυτά, λέγονται διάφορα σχετικά αστεία στην ε, Πολωνία, ότι πρέπει να πας πλέον για να βρει ζώο για, για κυνήγι. Ίσως θα πρέπει οι κυνηγοί να πιάνουν τα ζώα. Όχι μόνο τα κυνηγούν. Εντάξει, ίσως αστεία είναι αυτά που λέμε στην Πολωνία, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για το πώς θα αναπτύξουμε την τοπική παραγωγή. Θα πρέπει να υπάρχει ένας, ε, μια μικρή απόσταση ανάμεσα στον τόπο παραγωγής και στον τόπο κατανάλωσης και αγοράς μάλλον. Επίσης η τοπική αγορά ακόμα και αν δεν υπάρχει επισήμανση, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί ο, ο παραγωγός είναι γνωστός. Οι καταναλωτές πηγαίνουν σε αυτόν μία φορά τη εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα. υπάρχουν σχέσεις, τον ξέρουν. Φυσικά χρειαζόμαστε κάποια μορφή ε, επισήμανση στην αγορά, αλλά ελπίζω αυτό να με οδηγεί σε υπερβολικό διοικητικό άχθος. Αυτά και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Κομισιόν για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που σας υποβλήθηκαν. Κύριε Έρχαρτ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα. Η οι πρώτε ερωτήσεις. Τι σχεδιάζει στο επόμενο βήμα της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει. Όπως σωστά εξετέθη προηγούμενα, εμείς βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος ε, μιας νομοθετικής περίοδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την έκθεση, αυτές τις δύο εκθέσεις, τις συνέταξε από πλευράς της και τις δύο αυτές τις συνέταξε με την πρόθεση αφενός το θέμα αυτό όσο γινόταν καλύτερα μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να το αναλύσει και την τοπική, τα τοπικά προϊόντα γεωργίας και τις άμεσες πωλήσει και της νησιωτικής γεωργίας τα προϊόντα με διαφορετικές προσεγγίσεις που θα έδιναν διάφορες, διαφορετικές δυνατότητες. Πραγματικά ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδιαφέρεται γνήσια σε αυτά τα ερωτήματα να δώσει απαντήσεις. Σε αυτά τα θέματα τα οποία αναλύσαμε για την τοπική διάθεση προϊόντων, άμεσες πωλήσει να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα. Για παράδειγμα, στο ερώτημα κατά πόσον η σημερινή ελαστικότητα ή τα μέσα ελαστικότητας λειτουργούν καλά ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα στον τομέα της υγιεινής ή μπορούν να βελτιωθούν ή κάτι θα πρέπει να γίνει ενδεχόμενα ή όχι σχετικά. Αυτό ήταν ένα από τα μελήματα, ένα από τα σημαντικά βιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε και από την άλλη πλευρά στον τομέα της υγιεινής για παράδειγμα ποιες επιπτώσεις υπάρχουν στην ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνατότητες δηλαδή για μια τέτοια ελαστικότητα σε κάποια κράτη-μέλη αυτή η ελαστικότητα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για αυτά τα κράτη-μέλη σε άλλα όχι δεν δεν την εκμεταλλεύονται. Και μέσα σε αυτό το συσχετισμό να δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη και πώς αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη διάθεση αυτών των προϊόντων λιγότερο επιτυχώς ή περισσότερο επιτυχώς. Εδώ λοιπόν να δούμε το θέμα των ρυθμίσεων ελαστικότητας. Ποια, ποιες επιπτώσεις έχει η ελαστικότητα αυτή. Πρέπει να αλλάξει και αν ναι, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο. Και στη συνέχεια θα ήθελα δύο στοιχεία να προσθέσω, δύο επισημάνσεις να κάνω. Δηλαδή, το ότι εμείς είδαμε στις προκατακτικές εργασίες ε, για, σε αυτό το επίπεδο, είδαμε ότι με την ομάδα επαϊόντων που συγκαλέσαμε, συζητήσαμε σχετικά αναλυτικά και σε βάθος το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί ε, το πλαίσιο για την εμπορία άμεση εμπορία και διάθεση στην αγορά ενός τέτοιου γεωργικού προϊόντος. Με ποιους ορισμούς και ποια πλαίσια θα έπρεπε να γίνεται αυτό ώστε για τους αγοραστές, για τους καταναλωτές να υπάρχει ένα αξιόπιστο πλαίσιο δυνατότητας αγοράς ενός τέτοιου προϊόντος. Δηλαδή, συχνά θέσαμε το ερώτημα, τι αναμένει ο καταναλωτής όταν θέλει να αγοράσει ένα τέτοιο προϊόν από τον ίδιο τον εκμεταλλευτή, από τον ίδιο τον παραγωγό, με συγχωρείτε, τον ίδιο τον γεωργό. Τι πρέπει να κάνουμε. Συζητήσαμε με τους επαΐοντες ε, σχετικές πτυχές και αναλύσαμε το ότι για παράδειγμα για το κρέας, ότι θα πρέπει να είναι ζώα τα οποία εκτρέφονται και παχύνονται την ίδια τη γεωργική κτηνοτροφική εκμετάλλευση και δεν μεταφέρονται από αλλού. Και η σφαγή στο ίδιο το, στην ίδια την εκμετάλλευση δεν είναι εκείνο το οποίο αναμένει ο καταναλωτής, αλλά θα ήταν πολύ πιο σκόπιμο η σφαγή να γίνεται σε ένα κοντινό σφαγείο, για παράδειγμα σε ένα κοντινό χωριό, ώστε το, το κρέας από τον γεωργό από τη δική του παραγωγή να διατίθεται σε αυτό το σφαγείο και μετά στους καταναλωτές. Έχουμε σχεδόν ε, επακριβή αποτελέσματα για αυτή την ανάλυση των ενιών και των παραμέτρων τι θα πρέπει να γίνει με αυτά τα προϊόντα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Ένας άλλος τομέας που εξετάσαμε ποιος είναι. Είναι το ότι είπαμε ότι αν μια έννοια για την ετικετοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται και να προστατεύεται, για παράδειγμα ορεινό προϊόν, προϊόν ορεινής γεωργίας, για παράδειγμα μέσα στο πλαίσιο των ε, ενδείξεων προστασίας για τέτοια προϊόντα. Ποιο όνομα, ποιος χαρακτηρισμός ε, θα πρέπει εδώ να εξετάζεται ώστε να προστατεύεται ένα τέτοιο προϊόν. Και ακόμα δεν καταλήξαμε σε κάποιο ιδανικό, σε κάποια ιδανική πρόταση. Διότι είδαμε ότι είτε στα κράτη-μέλη ήδη υπάρχουν καλά λειτουργούντα συστήματα για τέτοιου είδους προϊόντα τοπικών ε, μονάδων εκμετάλλευσης και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τώρα μια ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινοτική, πανενωσιακή ρύθμιση, θα μπορούσαν να υπάρξουν τριβές και προβλήματα με καλώς λειτουργούσες ενδείξεις και στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα. Και αν δούμε την, από την άλλη πλευρά την έννοια φεγμιέ στη Γαλλία για την έννοια του γεωργοκτηνοτρόφου και που για κάποια προϊόντα ήδη κατοχυρώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, πρέπει να δούμε. Είναι ανάγκη να εισαχθούν κάποιες νέες πρακτικές και κάποια νέα πλαίσια. Μήπως αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα. Αν λοιπόν θέλουμε να κινηθούμε πανενοσιακά προς μια τέτοια κατεύθυνση, θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε εξειδικευμένα την επιλογή του προϊόντος, του χαρακτηρισμού του προϊόντος, ώστε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε χειροπιαστά μια πρόκληση την οποία πρέπει να επιλύσουμε και να είναι ας το πω έτσι πιασάρικη η έννοια ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να, να κατανοεί αμέσως εύληπτα να αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται και να μην δημιουργούνται συγχύσεις και προβλήματα ή τριβές με, άλλες, με άλλους ορισμούς ε, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να πω από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά μας ενδιαφέραν. Ιδιαίτερα να υπάρξει αναφορά σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία αναφέραμε στην έκθεσή μας που πρέπει να καλυφθούν υπό το πρίσμα των αναγκών των καταναλωτών. Και υπό τη σημερινή συγκυρία και πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει να υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες και ούτε έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια σχέδια να δημιουργήσει πανενοσιακές ε, κοινοτικές ρυθμίσεις για την άμεση διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊόντων, για παράδειγμα νησιωτικών προϊόντων. Κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το επανεξετάσει εν ευθέτω χρόνο, ανάλογα με τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν στις εκθέσεις της για αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, προσδοκάτε να σας υποβάλουν και άλλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Και στη συνέχεια θα μας προτείνετε το τι ποιο ήταν το επόμενο βήμα. Καλά δεν κατάλαβα. Α, ωραία. Θα επανέλθουμε πάντως ε, στο θέμα αυτό και στο μέλλον. Δεν βλέπω να υπάρχουν όμως άλλες ερωτήσεις. Οπότε τελειώσαμε αυτό το σημείο Σε διάταξη. Μισή. Οπότε, αυτό το τμήμα τη συνεδρίασης εδώ ολοκληρώθηκε. Στι 5.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ. Στι 5.30 γιατί τότε θα έρθουν ορισμένοι εξ αυτών. Οπότε για του υπόλοιπου, σα ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνουμε προ το παρόν και με μεγάλη μα χαρά Έχουμε όλους αυτούς τους ε, εκλεκτούς προσκαλισμένους σήμερα. Αύριο στις 9 ώρα θα συνεχίσουμε. Και παραλαμβάνει ο Πρόεδρος, σε 20 λεπτά στις 5 και μισή πρόκειται να συνδυάσουν οι συντονιστές.